Ladies and gentlemen, good afternoon. Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σημείο υπαρθμών 1, προφανώ έγκριση της ημερησιάς διάταξης. Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την αρχική πρόταση. Το υπαριθμόν 6 σημείο που αφορά την εξέταση των ανθρωπολογιών για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών και τη διαδικασία έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής αναβάλλεται. Το σημείο 26 που αφορά την ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου τη και του δικαιώματο παράσταση του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινική διαδικασία αναβάλλεται και αυτό. Υπάρχουν αντιρρήσει ή υποδείξει σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο το λόγο, επομένω ε, η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Σε ό,τι αφορά το σημείο ανακοινώσεις του Πρόεδρου δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και έτσι πηγαίνουμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών. Αν δεν λάβουμε κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου αφενός και της 10ης και 11ης Νοεμβρίου αφετέρου, θα θεωρήσουμε, επαναλαμβάνω, ότι εγκρίνονται. Σημείο 4. Καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Το λόγο έχει ο συγγητής ο κύριος Κέστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια από τα σημαντικά ζητήματα που άπτονται του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Καταρχήν κάποια προκαταρκτικά σχόλια. Νομίζω ότι εν γέννη υπάρχει συνένεση ως προς το ότι οι δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Συνεισφέρουν σημαντικά στην κοινωνική συνοχή. Τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα μπορούν να είναι ένας ε, πολύ καλός τρόπος ε, μεταξύ, για, την ε, προσέγγιση των πολιτών με τους διάφορους φορείς και τα διάφορα θεσμικά όργανα. Καλό θα ήταν να διασκεδάσουμε την καχυποψία των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με ορισμένες διαδικασίες. Θα έπρεπε επίσης ε, να δούμε και ένα άλλο στοιχείο ότι πολλές φορές έχουν ε, πάρει το ρόλο μιας διεθνούς οργάνωσης ε. ή μπορεί να δημιουργούν ε, να ασκούν επιρροή, να προσπαθούν να προβάλλουν κάποια θέματα. Υπάρχουν ιδρύματα που ζητούν, πραγματικά χάρη, ιδιωτικοποίηση, τα λοιπά Στη Γερμανία το Ίδρυμα Μπέτερμαν. Το σχέδιο κειμένου της Κομισιόν προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα. 8 Φεβρουαρίου χρονολογείται ε, το 2012 και όλα σε αυτή η πρόταση και έχει τα εξή βασικά σημεία. Το Ευρωπαϊκό Ιδρύμα είναι μια ακόμη νομική μορφή πέραν του εθνικού καταστατικού και αφορά ιδρύματα Δημόσιο συμφέροντος. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την άποψή του και θα πρέπει να λάβουμε επίση υπόψη μα ότι θα απαιτηθεί ανωνυμία στο Συμβούλιο για την έγκριση του κατεστατικού αυτού. Τα ευρωπαϊκά τρήματα έχουν προβλήματα όταν δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μια χώρες. Έχουν με ιδρύματα με διεθνωρικές δραστηριότητες. Εδώ όμως υπάρχουν διάφορα προσκόμματα φορολογικά, αστικού δικαίου. Όμως θέλουμε να ασκήσουν αυτές τις δραστηριότητες τους προς το δημόσιο συμφέρον τα ιδρύματα αυτά. και στα κράτη θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των διεθνών αλλοδαπών ιδρυμάτων. Όπως για τη Γερμανία, που θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ιδρύματα στην Γερμανία αυτά τα ξένα ιδρύματα. Υπάρχουν κάποια φορολογικά ωφέλη που δίνονται στα ιδρύματα αυτά. Η πρόταση της Κομισιόν είναι σε αυτό το καταστατικό να μπει σχετική διάταξη. Και άπαξ και εγκριθεί αυτό το καταστατικό, αυτό το καθεστώς, θα πάψει να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Και έτσι θα μπορούν να διεξάγουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες τα ιδρύματα αυτά. Ένα ίδρυμα με βάση αυτό το καθεστώς μπορεί να συσταθεί μόνο εφόσον στόχος του είναι το δημόσιο συμφέρον. Με βάση την πρόταση, ή οδήποτε κέρδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ακριβώς προς το δημόσιο συμφέρον. 25.000 ευρώ είναι το ελάστο κεφάλαιο και εκεί περιορίζεται και η ευθύνη σε αυτό το ποσό. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα πρέπει να δραστηριοποιείται σε διεθνέ επίπεδο και συγκεκριμένα πάνω από δύο κράτη-μέλη. Η έδρα, η βασική, μπορεί να είναι σε άλλο κράτος από αυτό στο οποίο ασκούνται δραστηριότητες. Δημιουργούνται όμως προβλήματα. Αν το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου αν δεν, δεν είναι σαφές ποια, ποιο δίκαιο πρέπει να τηρείται. Υπήρξε και μια ενδιάμεση έκθεση της κυρίας Ρέγκνερ Για το κατά πόσον διοικητική έδρα και καταχωρημένη έδρα πρέπει να είναι το ίδιο ή διαφορετικό. Επίσης λέγεται ότι θα πρέπει να εθαρρυνθεί ο εθελοντισμός. jede wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, ähm, Πρέπει να δούμε επίσης και το ενδεχόμενο να ασκούνται παράνομες δραστηριότητες, γιατί φυσικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό. Σε ποιο βαθμό λοιπόν τα διοικητικά γραφεία ή η εδρα θα πρέπει να είναι στο ίδιο στο, ή σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε. Και υπάρχει και ένα σχετικό θέμα, το πώς δηλαδή αυτό επηρεάζει τους εργαζομένους. Δεν έχει απαντηθεί το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις για τη δημιουργία των εργασιακών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Εργασιακού Συμβουλίου ή Επιτροπής Επιχείρησης, δεν προβλέπεται η συναπόφαση ή η συμμετοχή των εργαζομένων δηλαδή στις αποφάσεις. Για παράδειγμα στη Γερμανία τα εδρήματα εμπίπτουν ε, σε αυτό τον όρο περί συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Είπαμε τώρα το ελάχιστο κεφάλαιο, το ενεργητικό πρέπει να είναι 25.000. Στις 19 Νοεμβρίου του τρέχοντος το συζήτησε το θέμα η Κορεπέρ και τα περισσότερα κράτη-μέλη ήταν υπέρ του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Έδωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους. αλλά δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία, υπάρχει πλειοψηφία προ το παρόν. Απαιτείται όμως ομοφωνία, δεν ξέρω, ίσως έχουμε κάποιες ειδήσει μέσα στι επόμενε ημέρες. Κλείνοντα. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει η Συμβουλή, Okay. Επιτροπή να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις, ιδίως ό,τι αφορά το τι ισχύει σήμερα ε, για τα φορολογικά, για παράδειγμα, που είναι ένα σημαντικό θέμα ή κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Είναι σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσει με στόχο την επίτευξη ομοφωνίας. Εγώ νομίζω ότι εδώ ε, μπορούμε να συζητήσουμε παραπάνω το όλο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ντεγκράντες. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι δεν θα φτάσω γιατί καθυστέρησε η πτήση αλλά ευτυχώ κατάφερα όχι μόνο να είμαι εδώ τώρα, αλλά να ακούσω και τον εισηγητή. Το είχε ξαναπεί ε, και η κυρία Ρέγνερ ήταν τότε εισηγήτρια, εγώ ήμουν σκιώδης. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε αντιστρέψει τη σειρά και να μιλήσω ίσως πρώτα εγώ, γιατί ήθελα να σας πω το χρονικό μιας αποτυχίας. Στις 19 Νοεμβρίου στο Κορεπέρ 15 ψήφισαν, κράτη ψήφισαν υπέρ και 8 κατά. Δηλαδή, παρά τις αξιέπαινες ε, θετικές δράσεις της Ιταλικής Προεδρίας, ε, δεν ευωδόθηκε το θέμα, παρότι εμείς... Ε, είχαμε γνωμοδοτήσει ως ε, κοινοβούλιο, τα είπε και ο εισηγητής, και η Επιτροπή των Περιφερειών και η ΕΟΚΕ είχαν ε, εκφράσει τι τους και υπήρξαν και πάρα πολλές διαβουλεύσεις γύρω από την γενικευμένη πιστεύω ε, άποψη ότι πρέπει να έχουμε αυτό το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Είναι κρίμα που είχαμε 8 από τις 28 χώρες να λένε όχι σε αυτή την πρόταση που για μένα ήταν ε, τεκμηριωμένη. Βέβαια στη συζήτηση Προέκυψαν διαφωνίε, αυτό είναι άλλωστε φυσιολογικό. Νομίζω όμω ότι υπήρχε μεγάλη συνένεση στο Κοινοβούλιο. Γιατί η πλειοψηφία ήταν, θα έλεγα, συντριπτική στο Κοινοβούλιο κατά την ψηφοφορία. Υπήρχαν κάποια κριτήρια και νομίζω ότι συμφωνούσαμε όλοι ε, για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα και το καθεστώ τη. Θέλω να ακούσω το Συμβούλιο, πραγματικά καίγομαι, θα έλεγα, φλέγομαι, επιθυμία να ακούσω τι έχει να μα πει, για ποιο λόγο απέτυχε η διαδικασία εκεί. Ο εισηγητής μας μας υπενθύμησε κάποιες θέσεις. Θα σας πω και τι είχε γίνει όταν εγώ ήμουν σκιώδηση στη σοσιαλιστική ομάδα. Εγώ είχα, κάνει κάποιες, ε, είχα δώσει κάποιες προειδοποιήσεις. Γιατί υπήρχαν κάποια ζητήματα και μπορεί να μην μπορούσαν όλοι να δεχτούν εύκολα αυτή την πρόταση. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, κοινωνικο-οικονομικές, πάρα πολλές ανάγκες, οικονομικές, κοινωνικές υπάρχουν. Τα ιδρύματα έχουν ένα σημαντικό ρόλο, συνεπικουρούν ε, μαζί με τον ε, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει να είναι δημόσιο συμφέροντο, όπω είπα. Και είναι αποτελεσματικά εργαλεία αυτά τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Από την άλλη πλευρά όμω πρέπει να είναι και ελκυστικά. Αυτό το σύστημα με τις συμβατότητες στο Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά τις οικογένειες, δεν μου φάνηκε και έτσι και πολύ έξυπνο. Διότι ήθιστε οι μεγάλες και ισχυρές οικονομικά οικογένειες ε, να κάνουν δωρεές στην ε, κοινωνία υπό τη μορφή συγκρότηση δρυμάτων. Δίνουν πόρους λοιπόν για να μπορέσει να τους εκμεταλλευτεί η κοινωνία των πολιτών. Και πολλές φορές ε, η οικογένεια λαμβάνει τις ε, αρμοδιότητες με το το βέβαιο έλεγχο, γιατί δεν πρέπει να, είναι να, να λειτουργεί αυθαίρετα αυτό το Ίδρυμα, πρέπει όπως είπα να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Έχουμε το ζήτημα της εκπροσώπησης των εργαζομένων των Ιδρυμάτων. Ορισμένες φορές δεν είναι σωστό να υπάρχει υπερβολική ακαμψία για ατυπικά θα έλεγα ε, όργανα, φορείς. Εκεί πρέπει να έχουμε λίγο μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί αν έχουμε αυτό το άκαμπτο, π.χ. γερμανικό σύστημα της ε, συναπόφασης κατά κάποιο τρόπο, δεν θα μπορούν να επιτελέσουν αυτές τις δράσεις, ε, τις ωφέλιμες τα ιδρύματα. Και τα φορολογικά ζητήματα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα γιατί πρέπει σίγουρα να είναι ελκυστικά αυτά τα ιδρύματα, άρα πρέπει να έχουν κάποιες ίσω ε, ελαφρύσεις ή κάποια προνόμια. Θέλω να δω λοιπόν, ε, να ακούσω από το Συμβούλιο τι έγινε. Ακούσαμε ότι 15 χώρες ε, ετάχθησαν υπέρ και 8 κατά τη πρότασης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε, μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί αν συμφωνούμε όλοι σε κάτι, αυτό είναι ότι τα ευρωπαϊκά ιδρύματα μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που σέβεται και τη φορολόγια, την εθνική και την επικουρικότητα. Είναι προστέμενη αξία δηλαδή. Δεν ε, βλάπτει το status quo των κρατικών ιδρυμάτων. Δεν ξέρω γιατί το ανακόψαμε την πορεία του σκάφους αυτού που εμείς νόμιζαμε ότι ε, θα πήγαινε με ούριο άνεμο προς τα εμπρός. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Ε, thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Χαούτα. Thank you very much, Chair. <laughs> Um, I think there's... Δεν ε, υπάρχει αμφιβολία ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ε, το καθεστώς αυτό ε, υπέρ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Αλλά θα ήθελα να μου υποθεί γιατί τα οκτώ κράτη-μέλη εκφράζουν επιφύλαξη επί του θέματος και ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε το γιατί έτσι ώστε να εκπονήσουμε τελική πρόταση η οποία θα εγκριθεί. Έχω ορισμένα ερωτήματα που θα ήθελα να απαντηθούν από την Επιτροπή και τον εισηγητή. Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος ίσως διαφέρει από χώρα σε χώρα και θα ήθελα να ξέρω αν για παράδειγμα τα φορολογικά ευεργετήματα αυτών των ιδρυμάτων στη χώρα λειτουργίας με βάση την εργασία υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, εάν αυτό μπορούν να το προβάλλουν εύκολα, θα οδηγούσε και σε μία αρχή αμοιβαία αναγνώρισης, γιατί ίσως το δημόσιο συμφέρον να διαφέρει ανάλογα με το κράτος μέλος. Δεύτερον, διαβάζοντας τη γνωμοδότηση Επιτροπής Πολιτισμού, που συντάχθηκε 1,5 χρόνο πριν, θα ήθελα να μου υποθεί κατά πόσο αυτό που είπε η Επιτροπή Πολιτισμού, δηλαδή άνοιγμα, λογοδοσία, έλεγχος και ελάχιστες προδιαγραφές για την οικονομική δραστηριότητα, κατά πόσο αποτελεί μία εγγύηση που θα εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη μας σε αυτά τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Στην ομάδα μας συζητήσαμε και αναρωτιόμαστε πόσο θα μας πάρει μέχρι ότου αποφανθεί η Επιτροπή για μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί γνωρίζουμε ότι υπάρχει το θέμα ε, καταγραφή στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο. Όχι μόνο ε, για ε, θέματα φορολογικών ελαφρύνσεων και ευεργετημάτων. Αυτή η πρωτοβουλία δεν υπάρχει ακόμα επιτάπτητος. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε λοιπόν ε, να υποβάλουμε ένα ερώτημα προς το Συμβούλιο για την ανάγκη ε, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριο Φως. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, διάφορες πληροφορίες και συμφωνώ με τον κύριο Κέστερ, τον ενθαρρύνω μάλιστα να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα του κατακαιρματισμού της έδρας. Το είδαμε όπως και με τον, με τον κύριο Γκράντες με την μονοπρόσωπη εταιρεία, διότι σε ορισμένους τομείς οδηγεί σε ανεπιθύμητες ενέργειες. δεν πρόκειται για ε, φοροδιαφυγή, είτε πρόκειται για πλήσιμο βρώμικου χρήματος κλπ. Θέλουμε τη μορφή αυτή, αλλά θέλουμε και να λειτουργεί σωστά, χωρίς να ανοίγει παραθυράκια που υποτίθεται πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό και σας ενθαρρύνω και πάλι να εξετάσετε και τις ένομες συνέπειες της μορφής αυτής, ώστε να μπορέσουν να αποφευθούν ανεπιθύμητα φαινόμενα. Σωστή είναι βέβαια η ευκαμψία, όπως είπατε και εσείς και ο κύριος Δεγκράντες, και χρειάζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, να μην φτάσει όμως σε αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα να το εξετάσετε αυτό. Ευχαριστώ, Ράντιεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα υπάρχουν 110.000 ιδρύματα ε, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό και απασχολούν ένα εκατομμύριο πολίτες. Επίσης αυτά τα ιδρύματα ασχολούνται, έχουν μάλλον ένα πολύ ε, βαρύ φόρτο σε φορολογικά και διοικητικά ζητήματα και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν ε, για ε, πιο χρήσιμους σκοπούς. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσαν να μεταφερθούν πόροι, γνώσεις, και θα μπορούσαμε να μειώσουμε την ε, νομική ανασφάλεια που υπάρχει. Όμως έχει μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μία διαρκή απασχόληση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και ένας αποτελεσματικός έλεγχος. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δραστηριότητα των ιδρυμάτων αυτών. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε τα ιδρύματα να έχουν αυτό το μέσο που αναμένουν. Θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ισχύσει το νέο καθεστώς για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κνέφελ θα λάβει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής ή ο συνάδελφος. Θα αρχίσω εγώ. Και σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ιδιαίτερα από τον εισηγητή και την κυρία Ρέγνερ στο παρελθόν. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε ε, υποστήριξη από το Κοινοβούλιο επί του θέματος, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Και έτσι η Επιτροπή μπορεί να προ... προβάλλει μια πολύ καλή πρόταση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Ως προς το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρότασης έχουμε να κάνουμε με ιδρύματα δημόσιου συμφέροντος. Δηλαδή μιλάμε για εμπορικές δραστηριότητες. Μια μεγάλη επιχείρηση όπως το IKEA Έφνης αποκλείεται από αυτό το πλαίσιο. Μιλάμε για φιλανθρωπίες, δραστηριότητα των εκκλησιών και ούτω καθεξής, δημόσιο συμφέρον με λίγα λόγια. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσω σε επίπεδο λεπτομέρειας, αλλά σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Δελγκράντες, τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Μετά από τριετής διαπραγματεύσεις, 11 ομάδες εργασίας και 3 κορεπέρ, βρισκόμαστε στην κατάσταση όπου 8 κράτη-μέλη αντιτάσσονται σε αυτή την πρόταση, 5 θα ήθελαν αρκετές αλλαγές, ενώ οι, οι υπόλοιπε χώρες υποστηρίζουν θερμά ή μη την πρόταση. Υπάγεται στο άρθρο 352 της συνθήκης, άρα χρειάζεται ομοφωνία γιατί μιλάμε για το καθεστώς του Ιδρύματος. Ο κύριος Ντελγκράντε ρώτησε ε, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν, ε, δεν ξέρω εγώ ποια είναι τα προβλήματα ανακράτος. Δηλαδή κάνω το συνήγορο του διαβόλου εδώ από πλευράς Επιτροπής, αλλά οι περισσότερες ανησυχίες σχετίζονται με το ότι δεν βλέπουν ποια είναι η προστιθέμενη αξία της πρότασης. Δεν βλέπουν να υπάρχει προστιθέμενη αξία, διότι θα δημιουργούσε ένα νέο νομικό φόρουμ γι' αυτό. Το ευεργέτημα του καθεστώτος δεν θα υπερβεί το διοικητικό βάρος. Υπάρχει και το κόστος ελέγχου, η εγγραφή, ελάχιστο κεφάλαιο και ούτω καθεξής. Δηλαδή η προστιθέμενη αξία δεν φαίνεται να είναι σημαντική. Εμείς σε επίπεδο Επιτροπής αναγνωρίζουμε ότι τρία χρόνια μετά θα πρέπει να αποτιμήσουμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό είπαμε και στην Κορεπέρ δέκα μέρες πριν και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Όπως γνωρίζετε, στην Επιτροπή απασχολούμαστε με το πρόγραμμα εργασίας για το 2015 και αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που απαιτεί ομοφωνία και συνένεση του σώματος αυτού, καταλαβαίνετε τι εργασία σημαίνει. Οι διαπουλεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο επιτροπής και η Επιτροπή εργάζεται και επί ενός καταλόγου για να δούμε ποια ζητήματα πρέπει να αποσύρθουν, ποιοι φάκελοι πρέπει να αποσύρθουν. Είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά καθίστετε σαφές ότι αυτό το ζήτημα ίσως οδηγήσει σε μια τέτοια πρόταση. Βεβαίως θα ακολουθηθεί η σωστή η διαδικασία και θα τηρήσουμε και την ε, πολιτική διαδικασία. Ίσως να αφήσουμε τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση. Μία επιπρόσθετη παρατήρηση έχει ως εξής. Δεν υπάρχει μία πρόταση για μία Ευρωπαϊκή Ένωση Υποβλήθηκε μια πρόταση στη δεκαετία του 90 η οποία αποσύρθηκε ίσως ε, το θυμόσαστε στη DG Enterprise, το συζητήσαμε αυτό, αλλά οποιαδήποτε πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ομοφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει καταρχήν με το Ίδρυμα. Εάν απορριφθεί δεν θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ε, στο εγγύς μέλλον για το δίκαιο των επιχειρήσεων. Δεν ήθελα να είμαι αρνητικός και απεσιόδοξος, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κανένας άλλος από το Συμβούλιο δεν θέλει το λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο η συγγετής θέλει να κάνει μια τελική παρατήρηση, τελικές παρατηρήσεις. Μάλιστα. Θέλω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις συστάσεις σας καθώς επίσης και τη ρεαλιστική τοποθέτηση της Κομισιόν. Θα πρέπει να δούμε τώρα από την Νομική Επιτροπή ποιες ενδεχόμενα πρωτοβουλίες μπορούν να προκύψουν ώστε να ανοίξει πάλι ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα και να δοθεί και κάποια όθηση. Πρέπει να το συντονίσουμε όμως αυτό. Για τα ουσιώδη θέματα όπως ε, διάκριση μεταξύ διοίκησης και έδρας, αυτά είναι θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν, καθώς επίσης και θέματα συναπόφασης, βεβαίως με ευκαμψία ή ευελιξία για τους εργαζόμενους. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις παραπέρα διαβουλεύσεις. Όμως, ξαναλέω, πρέπει να δούμε κατά πόσο θα δραστηριοποιηθούμε ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αν θα ξεκινήσουμε κάποια πρωτοβουλία, για να δώσουμε κάποια όθηση και να πάρει μπρος πάλι η ε, υπόθεση. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Grandes και Χάουταλα επιθυμούν να επανέλθουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να είναι πιο συγκεκριμένη. Εγώ θα ήθελα όμως ε, να ακούσω πιο πολλές λεπτομέρειες ε, για το ποιο είναι που συνέβησαν αυτά που συνέβησαν στο Συμβούλιο. Μας είπατε ναι ότι 8 κράτη-μέλη ετέθησαν κατά, 5 θέλουν αλλαγές ε, και 3 είναι λίγο πιο ε, διαλλακτικοί θα μπορούσαν να δεχθούν ε, αλλαγές και έτσι να προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Νομίζω ότι είναι μια εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση πιστεύω συμφωνούμε όλοι ότι ε, η απότατη, ο απότατος στόχος αυτών των τερμάτων πρέπει να είναι το δημόσιο συμφέρον. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση. Έτσι όμως ερωτώ ποιο θα ήταν το νομικό μέσο που θα μας βγάλει από τα διέξοδο. Τολμώ να πω, να προτείνω, ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες, ε, μάλλον ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα των δυσκολιών με την ενισχυμένη συνεργασία. Και γιατί όχι, κάποιες φορές ε, από την τυπική νομική πλευρά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει λύση αν δεν υπάρχουν μεγάλες επί της αντιρρήσεις. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν θέλω να ασκήσω ε, κριτική στην Κομισιόν που ήταν φιδωλή ε, στις εξηγήσεις που μας έδωσε, το καταλαβαίνω. Ε, γιατί από την άλλη πλευρά δεν έρχεται εδώ να μας πει ότι φταίει αυτή, αφού φταίει το Συμβούλιο η Ιταλική Προεδρία ε, βέβαια το προσπάθησε. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Τώρα ποια είναι τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν σε αυτή την ε, ε, αρνητική ψήφο των 8 θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα. Τι αντιρρήσεις προέβαλαν τα κράτη-μέλη τα οποία τέθησαν κατά της πρότασης είναι κατηγορηματικές ε, αντιρρήσεις και ενστάσεις ή θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευέλικτοι ως κοινοβούλιο και να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Αυτά έχω να πω κύριε Πρόεδρε. Thank you, Mrs. Yeah, thank you. Ευχαριστώ κύριε Χαουτάλα. Θα μπορούσα να επαναλάβω τα όσα είπε ο κύριος Ντεγκράντες. Νομίζω ότι είναι κάπως ε, παράξενο το ότι συζητούμε για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός και δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιφυλάξεις των 8 χωρών στο Συμβούλιο. Δεν μπορεί οι θέσεις να είναι τόσο απόρριτες. Με ενοχλεί λοιπόν αυτό. Το γεγονό ότι όταν ρωτούμε η απάντηση που λαμβάνουμε είναι σιγή. Ο κ. Τεκράντες ε, σωστά ρώτησε, σωστά μάλλον πρότεινε, ότι μπορούν να είναι νέα χώρε οι οποίε θα προχωρήσουν στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Βέβαια, εγώ έλεγα το λόγο διότι έθεσα και συγκεκριμένες ερωτήσεις, ίσως να φαίνεται τα αγγλικά μου που δεν είναι τέλεια, αλλά δεν νομίζω ότι έλαβα απάντηση σχετικά, πόσο, σχετικά με το πόσο ποικίλει η έννοια του δημοσίου συμφέροντος στις ε, νομοθεσίες των χωρών μελών και ιδίως σε ό,τι αφορά τα ε, ωφελήματα της φορολογίας. Θα ήθελα να μάθω. Το ίδιο για, την, το θέμα της λογοδοσίας. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα ιδρύματα αυτά δεν θα καταλήξουν να γίνουν εργαλεία για το ξέβλημα του βρώμικου χρήματος. Ενώ τώρα συζητούμε σε ευρύτατο πλαίσιο την ε, απαγόρευση της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής κλπ. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σύντομα. Λυπούμε αν θεωρήσατε τις απαντήσεις μου επιφανειακές, πάλι δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό του Συμβουλίου, ούτε για λογαριασμό των 8 χωρών μελών. Θα σας εξηγήσω τι ακούσαμε. Θεωρούν ότι δεν είναι πεισμένες από την προστιθέμενη αξία της πρότασης. Αυτή είναι βασικά η γραμμή τους και θεωρούν επίσης ότι θα αυξηθεί το γραφειοκρατικό άκθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της φορολογίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για να διευκολύνει να αποφευθούν ε, αποκλήσεις φορολογίας μεταξύ των χωρών μελών. Αυτό ήταν σαν κόκκινο πανί για το Συμβούλιο. Ήδη από το 2013 οι μόνιμοι αντιπρόσωποι έλαβαν το ε, κεφάλαιο αυτό και το αφαίρεσαν από την πρόταση. Δεν λέει λοιπόν η πρόταση τίποτα πλέον για φορολογία σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Ίσως και για το λόγο που υπενήχθη κάποιος προηγουμένως για το ότι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή μπορεί να προκύψουν από κάποιες ε, αποκλήσεις που θα προκύψουν. Εμείς θεωρούσαμε πως όχι. Αλλά ολόκληρο αυτό το τμήμα του κειμένου έχει αφαιρεθεί. Αυτό βεβαίω μειώνει και την ίδια την την αξία τη προτάσεω. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία ακόμα υπέρ του τομέα αυτού, ώστε να θεωρεί ότι θέλει να προωθήσει την ε, πρόταση. Τώρα, το ενδεχόμενο κατακαιρματισμού των ευρών και οι σχετικέ παρενέργειε. Όλα αυτά, οι αλλαγέ επίση που έγιναν έγιναν με στόχο να μην υπάρχει δυνατότητα να διαχωρίζεται, να διαχωρίζονται οι έδρες, να υπάρχουν πλήρωνες έδρες δηλαδή του Ιδρύματος. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της ε, προτάσεως, μεταξύ αυτών δηλαδή περιλαμβάνεται και αυτό, και θεωρούμε ότι ο κίνδυνος της φοροαποφυγής κλπ. Έχουν, έχει μειωθεί σημαντικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος αυτού και λυπούμε βέβαια γι' αυτό. Έρχομαι στο 5 προσχώρηση της Αυστρίας και της Μάλτας στην σύμβαση της Χάγης του 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξοδίκων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις προς το σημείο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το λόγο έχει ο εισηγητής κ. Σουσπασκίχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εσείς κύριοι συνάδελφοι και κύριε συνάδελφοι, το θέμα μπορεί να παρουσιαστεί σύντομα. Το 1965, στις 15 Νοεμβρίου πιο συγκεκριμένα, υπογράφεται η Συμφωνία της Χόγης, που, Χάγης που επιτρέπει την επίδοση δικαστικών και εξωτικών εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σε άλλες υπογράφουσες χώρες, σε άλλες συμβαλόμενες χώρες. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επίδοση ρυθμίζεται σε άλλη συνθήκη που έχει υπογραφεί στις 2007. Το 2007 μάλλον, τον Νέμβριο πάλι του 2007. 26 χώρες μέλη της Ένωσης εφαρμόζουν ήδη την ε, σύμβαση αυτή. Τώρα, Αυστρία και Μάλτα επιθυμούν να προσχωρήσουν και αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το αποκριστικό δικαίωμα να χορηγεί εντολή στις ε, χώρες μέλη για να δεχθούν ή όχι την ε, προσχώρηση άλλων χωρών. Τέλος, στις 15 Νοεμβρίου 1965 όπως είπα εγκρίθηκε η σύμβαση της Χάγης και έχει αποδείξει την αξία της για την επίδοση δικαστικών ή εξωδικών εγγράφων. Όλες λοιπόν οι χώρες μέλη ενδιαφέρονται να έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο σύστημα επιδόσεως δικαστικών και εξωτικών εγγράφων. Προτείνεται λοιπόν η υποστήριξη, να χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξη στις αιτήσει αυτές της Μάλτας και της Αυστρίας. Ευχαριστώ. Έχετε κανένα σχόλιο, κύριε Ζιβιέφκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον εισηγητή εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος. Δηλώνουμε ικανοποιημένοι που επιθυμούν να ενταχθούν Μάλτα και Αυστρία στην Σύμβαση για την επίδοση δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική ρύθμιση για να εξασφαλιστεί η ομαλή απονομή της δικαιοσύνης και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποια χώρα μέλος θα μπορεί να παραμείνει απ' έξω. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και εγώ θεωρώ την προσχώρηση Μάλτας και Αυστρίας σημαντική. Άλλωστε, ανταποκρίνεται αυτό και στην δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 όταν έγινε ίδια μέλος της Σύμβασης της Χάγης. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει και σε τρίτες χώρες την προσχώρηση στις, στη σύμβαση αυτή. Επομένως, είναι απόλυτα φυσιολογικό οι δύο αυτές χώρες, Αυστρία και Μάλτα, που είναι ήδη μέλη της Ένωσης, να τα προσχωρήσουν στη σύμβαση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται λοιπόν να είναι αρκετά ξεκάθαρη η άποψη της ε, Επιτροπής Συνολικών Θεμάτων, όμως θα ψηφίσουμε όταν το Συμβούλιο θα ζητήσει την συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που θα γίνει σε μερικούς μήνες και όχι πιο πριν. Έχει αναβληθεί το υπαριθμόν 6, το υπαριθμόν 7, προσχώρηση του Μαρόκου στην Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της ε, διεθνούς απαγωγής τέκνων. Παρακαλώ κυρία Χάουταλα να λάβετε το λόγο εσείς ως εισηγήτρια. Έχω ήδη παρουσιάσει το σχέδιο εκθέσεως την προηγούμενη φορά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο παρά μόνο ότι επιτέλους το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατέληξε στο ότι πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν υπάρχει πλέον εμπόδιο. Ελπίζω ότι τα σχέδια εκθέσεων θα προχωρήσουν πλέον σε fast forward, διότι είναι προς το συμφέρον κυρίως των παιδιών που πέφτουν θύματα απαγωγής και μεταφέρονται σε αυτές τις τρίτες χώρες και των οικογενειών τους βέβαια. Υπάρχει μία πρόσθετη πληροφορία που θέλω να σας υποβάλω. Ρώτησα την νομική υπηρεσία την προηγούμενη φορά εάν υπάρχει κάποια κάποιο ενδεχόμενο το πεδίο εφαρμογής της συμβάσεως να επεκταθεί ώστε να περιλάβει και οι υποθέσεις παιδιών που θα έχουν προκύψει όταν θα τεθεί σε ισχύ, θα έχουν ήδη γίνει δηλαδή. Μου απάντησαν ότι δεν είναι δυνατό αυτό γιατί θα σήμαινε αναδρομική ισχύ. Ελπίζω λοιπόν ταχύτατα να προχωρήσει, αν υπάρχουν τροπολογίες θα τις εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Κανείς έχει σχόλια. Δεν βλέπω κανένα σχόλιο. Στην προκείμενη περίπτωση το, το Συμβούλιο έχει ζητήσει γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Άρα καλούμεθα να προβλέψουμε προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών η οποία θα είναι 8η Δεκεμβρίου ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον επόμενο το χρόνο, το Γενάρη. Αυτά για το 7. Um, for points number 8 and... Για τα 8 και 9 τώρα δεν είναι μαζί μας ο κύριος Καβαδά που είναι εισηγητής και αυτό βέβαια μας θέτει ενώπιον ένας προβλήματος διότι θα χρειαστεί τότε να αναβάλουμε τη συζήτηση των θεμάτων αυτών και άρα να προχωρήσουμε στο 11 και επόμενα τα οποία διεξάγονται τόσο και κλεισμένων των θυρών. Άρα θα παρακαλέσω όλες και όλους όσοι δεν έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Διάλειμμα 5 λεπτών.